δεν εγκεκριμένα. Ο κύριος Ντανιέλ Βαρέλα Κουάρες Καρπένια μετά από την παρέτησή του από τη θέση του Ευρωπαίου Βουλευτή ε, ε, ε ήδη ε, ισχύει λοιπόν αυτή η κατάσταση από τις 10 Μαρτίου, δηλαδή από χθε, και θα λάβουν γνώση οι αρμόδιες εθνικές αρχές. Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη